Επίσης θέλω να καλωσορίσουμε 25 νέους ε, από ένα εκδοτικό οίκο που έχουν προσκληθεί από την, κυρία, από την κυρία Ζαμπίνε Φεχάιεν. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Πολιτισμού. Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο ε, την έγκριση των πρακτικών της 22ης Ιουλίου. Το προηγούμενο σημείο ήταν η έγκριση της ημερήσιας διάταξης, την οποία εγκρίναμε και τώρα περνάμε ε, στα πρακτικά της 22ης Ιουλίου. Δεν έχουμε αντίρρηση, άρα προτείνω να εγκρίνουμε τα πρακτικά. des Vorsitzes Περνάμε στο σημείο 4, ανακοινώσει του Προέδρου. Να σα μιλήσω για τη διερμηνία στη σημερινή συνεδρίαση. Υπάρχει διερμηνία στα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσέχικα, ουγγρικά, λετονικά, πολωνικά, σλοβακικά, σλοβενικά, βουλγαρικά, ρουμανικά και κροατικά. Υπενθυμίζω ότι η σημερινή συνεδρίαση αναμεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Να περάσουμε τώρα στο θέμα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης ε, Εγκυκλοπαίδεια του 2019. Η κυρία Μελμπέρντε ζήτησε το λόγο για να μας ενημερώσει για μια εκδήλωση που γίνεται 11 και 12 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες με το όνομα European Encyclopedia Conference 2019. Δίνω το λόγο στην κυρία Μελμπέντε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τον Οκτώβριο θα γίνει η Ευρωπαϊκή Μέρα των Εγκυκλοπηδιών. Ε, και θα υπάρχουν εκπρόσωποι από τουλάχιστον 16 χώρες. καθώς επίσης ε, και ε, εκπροσώπηση από το Τμήμα Ερευνών του Κοινοβουλίου θα είναι η πρώτη φορά που εγκυκλοπαίδειες από όλες τις χώρες αλλά και από τις Ευρωπαϊκές Ένωση, αλλά και από την Βόρεια Αμερική θα μιλήσουν ε, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, προκλήσεις του μέλλοντος κλπ. Θα προκύψουν πολλές ερωτήσεις ε, και επιχειρήματα σχετικά με τον λόγο για τον οποίο χρειαζόμαστε τις εγκυκλοπαίδειες ε, στην, τον αιώνα των ε, πληροφοριών ε, του διαδικτύου και να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ε, που πιστεύουν ότι ε, στην περίοδο ακριβώς των fake news, ψευδών ειδήσεων ε, κλπ. χρειαζόμαστε τις εγκυκλοπαίδειες με την έννοια ότι οι εμπειρογνώμονες χρειάζονται επιβεβαιωμένες πληροφορίες και πληροφορίες τις οποίες να, οι οποίες να έχουν προετοιμαστεί από οι δήμονες και επομένως να είναι αξιόπιστες για τους ερευνητές. Τα τελευταία χρόνια η Υπηρεσία Μελετών του Κοινοβουλίου έχει σε βάθος μελετήσει την κατάσταση των πραγμάτων σχετικά ε, με τις επιγραμμικές εγκυκλοπαίδειες. Θα ήθελα να πω επίσης ότι οι οργανωτές μου ζήτησαν να οργανώσω και μία μικρή εκδήλωση ε, για τους ε, κοινοβουλευτικούς ε, και για τους βουλευτές λοιπόν και γι' αυτό λοιπόν θα έρθω σε επαφή μαζί σας έτσι ώστε να κάνουμε αυτήν την εκδήλωση την 9η Οκτωβρίου και θα χαρώ πολύ ε, να δω συναδέλφους και σε αυτήν την ε, μικρή εκδήλωση αλλά και μετά ε, στις εργασίες αυτής της συνάντησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Μελμπέντε και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο για την Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Έχουμε μια συζήτηση για την πολυγλωσσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, στις 26 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Στην τελευταία συνάντηση των συντονιστών αποφασίσαμε να οργανώσουμε μία συζήτηση για το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας. Εμπνευστήκαμε από την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών το 2001 και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, αποφάσισαν ε, κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου να εορτάζεται η Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Με την αφορμή αυτή οργανώνονται εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη οι οποίες ε, παρακινούν τους πολίτες ε, να ενδιαφερθούν για τις ε, γλώσσες που ομιλούνται στην Ευρώπη και να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Η κοινή διακήρυξη του 2001 παραμένει επίκαιρη. Σύμφωνα με τη διακήρυξη αυτή, όλοι κερδίζουν ε, τη δυνατότητα να υποφεληθούν από την πολιτιστική και οικονομική ε, πολυγλωσία, από τα πλεονεκτήματα της γνώσης ξένων γλωσσών. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών ε, συνεισφέρει σε μεγαλύτερη ανεκτικότητα και καλύτερη κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων με διαφορετικά γλωσσικά και πολιτιστικά υπόβαθρα. Στη σημερινή μα συζήτηση θα ήθελα να καλωσορίσω δύο προσκεκλημένους. Την κυρία Όλγα Λόμοβα, ε, ειδική για κινέζικη λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα και τον κύριο Μίχαηλ Τόιτς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μας μιλήσουν για την πολυγλωσία και για την εκμάθηση γλωσσών. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θα δώσω το λόγο για 10 λεπτά στην κυρία Λομόβα που θα μας μιλήσει για τη σχέση γλώσσας και πολιτισμού. Good morning ε, Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ που με καλέσατε για, για, με την ευκαιρία αυτής της συνάντησης. Πριν κάνω παρατηρήσεις ε, για την ε, κουλτούρα και την γλώσσα. Να σας πω ότι ε, στο Πανεπιστήμιό μας στην Πράγα ε, θα γιορτάσουμε την ημέρα των γλωσσών με μια πλήρη ημέρα δραστηριοτήτων όπου θα παρουσιάσουμε όλες τις γλώσσες που μπορεί κανείς να μάθει είτε στο Πανεπιστήμιό μας είτε σε άλλα Ινστιτούτα στην Πράγα. Θα προσπαθήσω να τις καταμετρήσω. Είναι πάνω από 40 40 ε, γλώσσες λοιπόν, όχι μόνο ευρωπαϊκές αλλά και ασιατικές. Ε, έχουμε προχωρήσει πολύ και μονάχα στις αφρικανικές γλώσσες υστερούμε και προσπαθούμε να ε, κερδίσουμε αυτό το, αυτό το έλλειμμα. Ε, πραγματικά ε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ε, συνολικά, να δούμε από κοινού το θέμα του πολιτισμού, της κουλτούρας και της γλώσσας. Και οι, και οι φοιτητές μας επίσης διαπιστώνουμε ότι θέλουν πολύ γρήγορα να μάθουν μια άλλη γλώσσα και μερικές φορές η προσαρμογή σε αυτήν την ταχύτητα της σύγχρονης ζωής μας κάνει να ξεχνούμε ότι η διαδικασία της μετάφρασης από μια, χώρα, από μια γλώσσα συγγνώμη, σε μια άλλη δεν ε, είναι μια απλή μεταγραφή εκφράσεων και ε, λέξεων είναι και η μετάδοση κάποιων πολιτιστικών στοιχείων ε, και μερικές φορές ε, μπορεί ακόμα και να ε, σχεδιάζει τον ίδιο τον πολιτισμό, την ίδια την κουλτούρα. Στην ουσία δηλαδή μέσω της μετάφρασης παρουσιάζουμε έναν ολόκληρο κόσμο. Διδάσκω πολλά χρόνια και μεταφράζω πολλά χρόνια. Έχω συχνά ε, υπάρξει ομιλήτρια σε πολλές γλώσσες, αλλά βεβαίως ε, επαγγελματικά ασχολούμαι με την κινέζικη. Έχω μεγάλη εμπειρία λοιπόν ε, και από την καθημερινή μεγάλη μου αυτή εμπειρία οφείλω να υπογραμμίσω ότι η εκμάθηση της γλώσσας συνεπάγεται και εκμάθηση του πολιτισμού. Σημαίνει ότι γίνεσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος όταν ε, αλλάζεις γλώσσα, στην ουσία πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να ε, χρησιμοποιήσεις ε, κάποιους κώδικες και αλλάζεις και σαν άνθρωπος. Πολιτιστικά λοιπόν γίνεσαι άλλος όταν αλλάζεις γλώσσα και η κατανόηση που έχεις ε, για τον κόσμο στην ουσία αντικατοπτρίζει ή μάλλον μορφώνεται, ε, διαμορφώνεται ε, ανάλογα με τη γλώσσα που ε, μιλάς. Βεβαίως θα πρέπει κανείς να ξέρει τη γλώσσα, να ζει τη γλώσσα, να έχει ενσυναίσθηση όσον αφορά την άλλη γλώσσα. Θα πρέπει να έχει πολιτιστική και γλωσσική ενσυναίσθηση. Ε, και τότε ενδεχομένως να αρχίσει να κατανοεί καλύτερα και τις προηγούμενες εμπειρίες του. Στα τσέχικα, όπως και σε άλλες γλώσσες, ε, λέμε ότι όσες γλώσσες μαθαίνεις, τόσες... Ε, experience it very much. Τόσες ζωές ζεις ή τόσα διαφορετικά, τόσα διαφορετικά άτομα μπορείς να είσαι. Ναι, έχουμε εδώ ένα παράδειγμα, το παράδειγμα της λέξης culture. Now I see it. <laughs> okay. Yeah. Uh, I thought, okay, let's, let's try. Ωραία. Είπα να δούμε λοιπόν την λέξη culture και ήλεγξα την ε, λέξη αυτή σε τέσσερους, ε, σε τέσσερα λεξικά. και βλέποντας τον ορισμό το, της λέξης ε, culture που είναι αρκετά περίπλοκος, προσπάθησα να δώσω και κάποια παραδείγματα από την καθημερινή χρήση που διαφέρουν από τις έννοιες που βλέπουμε ε, στα λεξικά. Πρώτα άνοιξα το Oxford Dictionary. Δίνει πολλούς ε, ορισμούς βέβαια, αλλά μπορούμε συνοπτικά να πούμε ότι ο ορισμός υπογραμμίζει κυρίως την κοινωνική ύπαρξη, την κοινωνία, τις κοινωνικές δομές, τα κοινωνικά ήθη και έθιμα ως δημιουργούς πολιτισμού. Επίσης ε, γίνεται αναφορά σε λογοτεχνία κλπ. Και πάντα ε, στα κοινωνικά δίκτυα. Αν δούμε τώρα λίγο το τσέχικο λεξικό, ε, με έκπληξη διαπιστώνομαι ότι ε, έχουμε περίπου τους ίδιους ορισμούς. Ακόμα πιο απλά θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι τόσοι πολλοί και παρόλα αυτά η κατανόηση ε, του πολιτισμού, της κουλτούρας σχετίζεται ε, με το πώς βλέπει κανείς αυτή την κουλτούρα. Ας πούμε στην ε, περίπτωση της Τσεχίας η επιστήμη έρχεται πρώτη σαν παράδειγμα από, το, από την λογοτεχνία. Έχουμε και το Merriam Webster. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ε αλλά ε, να πω ότι έχει και κάποιες διαφορετικές έννοιες από το ε, Oxford Dictionary, ε, πράγμα που δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί ο ορισμός ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Έχουμε και την άλλη άποψη ε, όπου αναφέρονται εξειδικευμένες έννοιες ε, και κάποιες ε, έννοιες που λείπουν τελείως από, την Ευρωπα... από τους ευρωπαϊκούς ορισμούς. Στην κινέζικη πλευρά, ας πούμε, αναφέρεται ως culture και η, ικανότητα συγγραφής ή η ικανότητα να κινείσαι σε κάποια περιβάλλοντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά των ορισμών σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας γλώσσα. Ε, δεν ξέρω τι λένε οι... Ε, ε αυτοί που έχουν αγγλική μητρική γλώσσα, αλλά μπορώ να σας πω ότι οι Τσέχοι όταν αναφέρονται σε culture, ε, σε πολιτισμό, αναφέρονται στην τέχνη, ενδεχομένως την ψυχαγωγία. Όταν ήμουν νέα βέβαια η ψυχαγωγία δεν αποτελούσε μέρος του πολιτισμού, τώρα ναι. Ε, ή όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα τα οποία ε, είναι, χρησιμοποιούνται πολύ και προβάλλονται πολύ τώρα. Ενώ στα κινέζικα μπορεί κανείς να εκπλαγεί βλέποντας ότι υπάρχει μία ε, ένας ορισμός, μια έννοια η οποία συνδέεται με την, τον πολιτισμό της ε, οικογένειας, ε, ε, δηλαδή κάτι το οποίο σχετίζεται με την εκδήλωση ειδικών εθήμων και στο, αγγλικό λεξικό, στο κινέζικο συγγνώμη, λεξικό διαβάζουμε σε σχέση με τα ρούχα, με την κόμωση, με το φαγητό, με τη συμπεριφορά ενώ αυτά τα στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνονται στον δικό μας ορισμό της ε, κουλτούρας. Βλέπουμε επίσης ότι η γλώσσα μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε κάθε φορά τη διαφορετική πραγματικότητα και καταβάλλονται προσπάθειες ε, από την ε, κοινωνία έτσι ώστε με κάποιο τρόπο να ε, καθορίσει κάποια στοιχεία, ε, να περιγράψει αποτελεσματικά τις, τις λέξεις μας, που ενδεχομένως στην επίσημη εκδοχή να διαφέρουν από την κατανόηση, την καθημερινή ας πούμε της ε, γλώσσας. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε εδώ ότι η γλώσσα έχει μεγάλη ευελιξία ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί το ίδιο το περιβάλλον αυθόρμητα δημιουργεί ε, νέες ε, αντιλήψεις ή, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να περιορίσει ε, τις έννοιες οι οποίες δεν έχουν πλέον χρήση. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκη ε, περίπλοκη η διασύνδεση της γλώσσας και του περιβάλλοντος εντός του οποίου ε, η γλώσσα δημιουργείται ή διαμορφώνεται. Τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε και να χαιρόμαστε ε, με την ποικιλομορφία των γλωσσών ε, είναι σημαντικό όχι μόνο να, προστατέψουμε τη δικιά μας κατανόηση ε, απέναντι στους άλλους, αλλά να καταλάβουμε καλύτερα τους άλλους μέσα από τη γλώσσα και με τον τρόπο αυτό ε, σίγουρα θα κατανοήσουμε και εμείς οι ίδιοι καλύτερα το δικό μας πολιτισμό, τη δικιά μας κουλτούρα. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια να κατανοήσουμε και να γνωστοποιήσουμε την ε, διαφορετικότητα. Αυτά ήθελα να σας πω μέσα από αυτές τις ε, λίγες παρατηρήσεις. Ε, ναι, και θα μπορούσα να τα είχα πει στα τσέχικα. Τώρα το συνειδητοποιώ αυτό. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λομόβα. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Τόιτς, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα μας κάνει μια παρουσίαση για τα μαθήματα γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Τότσο, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φραντς. Θα χρησιμοποιήσω το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου για να σας αναφέρω τις σημαντικότερες προκλήσεις που τίθεται και την πολιτική μας. Αναφέρατε την Ευρωπαϊκή Μέρα γλωσσών. Αν σας ενδιαφέρουν οι εκδηλώσεις που γίνονται στην κάθε χώρα, δείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής ή του Συμβουλίου της Ευρώπης και υπάρχουν αυτά τα θέματα για τα μαθήματα γλωσσών και η ίδια η Επιτροπή έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάνω από 100 εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή μέρα γλωσσών. Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στη σελίδα μας. Μιλήσαμε για τις διάφορες προκλήσεις. Ο στόχος μας είναι να μαθαίνονται ε, άλλες δύο γλώσσες παράλληλα με τη μητρική γλώσσα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος για την εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας, πολύ σημαντική η πρόοδος. Βλέπετε την εξέλιξη από το 2003 μέχρι το 2016. Το δίκτυο Ευρυδίκη έχει παράγει αυτά τα αποτελέσματα η πρώτη ξένη γλώσσα αρχίζει να διδάσκεται νωρίτερα και πολύ πιο συχνά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Είναι πολύ καλή λοιπόν η εξέλιξη για την εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας. Είναι λίγο διαφορετική η εικόνα για την εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας. Εδώ δεν, δεν φαίνονται τόσο θετικά τα αποτελέσματα. Πάλι η εξέλιξη από το 2003 στο 2016 δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος στο πώς διδάσκεται η δεύτερη ξένη γλώσσα, στο πόσο νωρίς ξεκινάει η εκμάθηση. Βλέπετε σε ποιες χώρες ξεκινάει από τα 11 ε, και μετά ή από τα 12, 13, 14. Είδαμε ότι υπάρχει πρόοδος λοιπόν στην εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας, αλλά για τη δεύτερη ξένη γλώσσα δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόοδος. Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης πάλι υπάρχουν ακόμη πιο σημαντικές προκλήσεις. Έχουμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη ποιο είναι ο στόχο. Ο στόχο είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών για όλου. Δηλαδή και αυτοί που έχουν την ε, εκπαίδευση του κλασικού ε, γυμνασίου και λυκείου, αλλά και για την επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει ε, οι μαθητές να μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα. Εδώ βλέπετε τις γλώσσες οι οποίες διδάσκονται περισσότερο. Δεν θα σας εκπλήσουν τα αποτελέσματα. Τα αγγλικά είναι η γλώσσα που έχει ε, το μεγαλύτερο ποσοστό εκμάθησης. Και ακολουθούν τα γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ρωσικά και ιταλικά. Τα αγγλικά όμως βλέπετε σαφώς δεσπόζουν σε αυτό το πεδίο. Έχουμε συζητήσει και το θέμα των μαθημάτων τα οποία προσφέρονται σε κάθε γλώσσα. Οι μαθητές συμμετέχουν σε μαθήματα εκμάθησης γλωσσών, αλλά δεν είναι πάντοτε εξίσου θετικά τα αποτελέσματα. Μπορεί να διδάσκονται μια ξένη γλώσσα, αλλά δεν είναι τόσο καλές οι ικανότητές τους ε, στο τέλος των μαθημάτων. Και εδώ έχουμε μία ε, καταγραφή των αποτελεσμάτων της ε, διδασκαλίας γλωσσών. Ποιο είναι το αποτέλεσμα στο οποίο έχουν φτάσει οι μαθητές μετά από ε, κάποια χρόνια διδασκαλίας της γλώσσας. Βλέπετε ποιοι είναι σε ενδιάμεσο, προ μεσαίο επίπεδο ή στοιχειώδες ή επίπεδο αρχαρίων. Για να φτάσουν τα παιδιά μετά από κάποια χρόνια σε επίπεδο Β1, Β2. Είναι κάθε φορά διαφορετικό το επίπεδο και βλέπετε και στο slide αυτό ότι είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα. Είδαμε ότι με την πρώτη γλώσσα, ε, όπου είναι και πιο υψηλά τα αποτελέσματα, τα αγγλικά είναι de facto η πρώτη ξένη γλώσσα. Η δεύτερη ξένη γλώσσα δεν ε, είναι υποχρεωτική παντού. Είδαμε ότι οι πρώτες γλώσσες είναι τα αγγλικά, γαλλικά, ε, ισπανικά, γερμανικά. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές γλώσσες στην Ευρώπη. Η πολυγλωσσία είναι σημαντική και δεν μιλάμε μόνο για αγγλικά, γαλλικά, ε, ισπανικά. Μπορεί να μάθουν τα παιδιά και πορτογαλικά και βουλγαρικά και λιθουανικά. Αυτό θα σήμαινε πραγματική πολυγλωσσία. Συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα και μετά από την ανάλυση μας θέλουμε να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους έχουμε για την πολυγλωσία. Στην άτυπη διάσκεψη κοινωνικών θεμάτων στο Γκέτεμπορκ πριν από δύο χρόνια συζητήθηκε αυτό το θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. με συμμετοχή και του Κοινοβουλίου για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα συστήματα εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευση. Δεν έχουμε ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση, αλλά ένα χώρο για την ε, εκπαίδευση. Και σημαντικό είναι ε, να υπάρχει κινητικότητα για να ε, και να μπορούν οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι στην Ευρώπη να έχουν τις γνώσεις των γλωσσών που απαιτούνται για την ε, καθημερινή τους επαγγελματική απασχόληση. Και θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, να υπάρχει αλληλοϊποστήριξη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται εκεί όπου υπάρχει αρμοδιότητα, αλλά θέλουμε ε, να διευκολύνονται οι αποφάσεις υπέρ της πολυγλωσσίας. ως στόχο είχαμε θέσει την εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών για να μπορούν περισσότερο οι νέοι στην Ευρώπη να μιλούν δύο επιπλέον γλώσσες εκτός από τη μητρική τους γλώσσα. Θέλουμε να δώσουμε μια νέα όθηση για να μπορέσει να επιτευχθεί καλύτερα αυτός ο στόχος. Και γι' αυτό δόθηκε και μια σύσταση με στόχους για την επίτευξη αυτής της σύστασης. Είναι σημαντική η γλώσσα στην οποία διδάσκεται κάποιο μάθημα, άρα με τη διδασκαλία των μαθημάτων σε διαφορετικές γλώσσες μπορεί να, γίνει, μπορεί να γίνεται καλύτερη εκμάθηση και να χρησιμοποιείται η πρώτη γλώσσα, η γλώσσα της σχολικής εκπαίδευσης με απόλυτα καλή γνώση, ενώ παράλληλα μια δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιείται σε επαρκές, επαρκώς καλό επίπεδο για κοινωνικούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Και μια τρίτη γλώσσα θα είναι μια γλώσσα στην οποία ο κάθε μαθητής, ο κάθε πολίτης θα έχει ένα επαρκή βαθμό γνώσης. Είμαστε υπερήφανοι για την ε, πολιτισμική πολυμορφία και το ερώτημα που τίθεται είναι τι κάνουμε χωρίς αγγλικά. Είναι τα αγγλικά μια γλώσσα χωρίς την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι μια γλώσσα στην οποία ε, επικοινωνούν οι περισσότεροι πολίτες και είναι σημαντικό να μαθαίνουν ε, οι μαθητές, οι πολίτες και μια δεύτερη γλώσσα. Πώς θα επιτύχουμε τώρα τους στόχους μας. Το συζητήσαμε με τους εμπειρογνώμονες και στο Συμβούλιο. Θα πρέπει το μάθημα να γίνεται με μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τις γλώσσες. Το μάθημα της γλώσσας δηλαδή να είναι σωστά ενταγμένο στο σχολικό πρόγραμμα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και την κινητικότητα και των διδασκομένων και των διδασκόντων. Να εξετάσουμε τρόπους ε, ε, επικύρωσης και άλλων μικρών γλωσσών. Εγώ σπούδασα στο Αμβούργο και για το απολυτήριο του σχολείου, για το απολυτήριο του Λυκείου, θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει μια δεύτερη ξένη γλώσσα, βουλγαρικά παραδείγματο χάρη, για να μπορέσει να συνεισφέρει στο βαθμό του απολυτηρίου. Η κατάρτιση των διδασκόντων είναι σημαντική. Και στο πλαίσιο των σπουδών τους, οι διδάσκοντες είναι καλό να περνάνε και κάποιες περιόδους ε, στο εξωτερικό. Είναι κάτι που δεν γίνεται υποχρεωτικά παντού. Είναι πολλοί πόροι οι οποίοι διατίθενται για τους ε, εκπαιδευτικούς, μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν. Βλέπετε ε, στην οθόνη πολλά παραδείγματα. Υπάρχει πολύ υλικό, υπάρχει το πρόγραμμα Erasmus, το Erasmus Plus. Ένα πρόγραμμα το οποίο σας έχει απασχολήσει και εδώ, τους τελευταίους μήνες νομίζω ασχοληθήκατε πολύ με το Erasmus Plus. Είναι ένα πρόγραμμα που προωθεί την κινητικότητα, τη συνεργασία, ένα σημαντικό στόχος που παίζει σημαντικό ρόλο για τη ζωή των πολιτών στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τόιτς για την ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Τώρα έχουμε χρόνο για να δώσουμε δύο λεπτά στον κάθε ομιλητή για ερωτήσεις. Θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία ping-pong. Η μία ερώτηση θα ακολουθείτε από απάντηση. Όταν θέτετε μια ερώτηση, να μας λέτε σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας για να μπορεί να απαντήσει. Εμείς θα κρατάμε κατάλογο ομιλητών Και καταρχήν δίνω το λόγο στους συντονιστές. Ξεκινώντας με την κυρία Ζιόντροβα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσω τσεχικά να ευχαριστήσω την κυρία Λόμοβα για την παρέμβασή της που μίλησε για την σχέση μεταξύ γλώσσας και πολιτισμού. Δεν θέλω να σπαταλήσω πολύ χρόνο, θέλω να θέσουν ερωτήματα φαντάζομαι οι συνάδελφοι για την εμπειρία της ε, κυρίας ε, ε, με την εκμάθηση των Κινέζικων. Ε, εάν θέλει κάποιος να μάθει Κινέζικα, εγώ θα ήθελα να ξέρω πόσος χρόνος χρειάζεται. Και ένα ερώτημα προς τον κύριο Ντόιτς. Δεν συμφωνώ και τόσο με αυτή την αντίληψη σύμφωνα με την οποία όλοι οι μαθητές 14 ε, με 15 ετών πρέπει να μάθουν μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Στην Τσεχία είναι υποχρεωτικό όντω. και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ούτε την πρώτη ξένη γλώσσα δεν μαθαίνουν καλά. Είναι πιο σημαντική η ποιότητα από την ποσότητα λοιπόν μία καλή ξένη γλώσσα να μαθαίνουν τα παιδιά και κάποια παιδιά που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και που μπορούν να το κάνουν, να έχουν τη δυνατότητα να μάθουν μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Το να γίνεται αυτό όμως υποχρεωτικά, όπως ισχύει επαναλαμβάνω τώρα στην Τσεχία, και μάλιστα δίνεται εντύπωση ότι το επιβάλλει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει στην πραγματικότητα ότι τα παιδιά δεν μιλούν καλά την πρώτη ξένη γλώσσα τους. Κάποια παιδιά δεν έχουν τόση έφεση στις γλώσσες, δυσκολεύονται ήδη με τα αγγλικά, δεν τα μαθαίνουν καλά, αναγκάζονται να μάθουν και μια δεύτερη γλώσσα, τα γερμανικά, φερρυπίν, και τελικά δεν μιλούν καμία ξένη γλώσσα καλά. Είναι λοιπόν σημαντικό να μάθει κανείς καλά μια ξένη γλώσσα και η δεύτερη πρέπει να είναι ε, δυνητικό αυτό για τα παιδιά που ενδιαφέρονται. Μπορεί να φορά τα μισά παιδιά. Το λέω αυτό και ως ε, πρώην ε, καθηγήτρια γαλλικών. Είμαι υπέρ της προώθησης των γαλλικών και της εκμάθησής τους, αλλά το βασικό είναι τα παιδιά να μπορούν να μάθουν καλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Από τη δική μου εμπειρία πάντως ε, νομίζω ότι το πρόβλημα ε, σχετίζεται με τη δεύτερη παρατηρήσή σας. Ε, ε, πρέπει να δούμε τι γίνεται στην πραγματικότητα. Πώς δηλαδή κανείς στην γλώσσα αυτή ε, μπορεί να βελτιωθεί. Τα κινέζικα, παραδείγματος χάρη, είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα προς εκμάθηση. Διότι για να μπορέσει κάποιος να ζήσει την πραγματικότητα μιας χώρας, της Κίνας στην προηγούμενη περίπτωση, είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι που βοηθάει να ζήσει κανείς την πραγματικότητα της χώρας. Βεβαίως ε, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο ακόμα. Η γιαγιά μου γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα με πολύ βασική εκπαίδευση. Μιλούσε όμως δύο γλώσσες διότι ζούσε σε έναν ε, δίγλωσσο κόσμο. Πιστεύω λοιπόν το να μάθει κάποιος τη γλώσσα εντάξει ο καθένας ε, βεβαίως έχει το ταλέντο του, έχει την έφεση που έχει αλλά όταν κάποιος εκτίθεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, δεν είναι πια θέμα έφεση και ταλέντου. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να μάθουμε μία γλώσσα όταν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που, υποχρεούμαστε να την χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Ναι, η κυρία Σιόντροβα έθεσε ένα σημαντικό θέμα. έχει δώσει τη γνώμη του και το Συμβούλιο. Ε, εμείς ως Επιτροπή πιστεύουμε ότι ε, είναι καλό να διδάσκεται μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Η πρώτη ξένη γλώσσα εξορισμού είναι τα αγγλικά. Και είναι μεγάλος ο πλούτος των γλωσσών στην Ευρώπη. Όταν θέλει κανείς να γνωρίσει ε, ε, μια χώρα, τη Σλοβακία, την Πορτογαλία, οποιαδήποτε, μπορεί κανείς με τα αγγλικά να τα καταλάβει, αλλά η γλώσσα βοηθάει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία να μαθαίνουν τα παιδιά και μια δεύτερη ξένη γλώσσα. μέσω της εκμάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας δεν φύγεται η εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας. Δεν θα συμφωνούσα απαραίτητο με αυτή την εκτίμηση. Και το επίπεδο το οποίο αναφέραμε είναι σημαντικό ότι η πρώτη ξένη γλώσσα είναι σημαντική για να μπορεί κανείς να δουλέψει ή να σπουδάσει στη χώρα της οποίας τη γλώσσα μαθαίνει. Η δεύτερη ξένη γλώσσα απαιτεί χαμηλότερες ικανότητες για να μπορεί απλώς να επικοινωνήσει κανείς. Είναι ένα θέμα πάντως πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Κάμερα Πέτχα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ δεν συμφωνώ με τη συνάδελφο. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξεκινά κανείς όσο το δυνατόν νωρίτερα. Γιατί ξέρουμε ότι τα μικρά παιδιά μαθαίνουν πολύ γρήγορα τις γλώσσες. Ήδη από τον παιδικό σταθμό, μέσω του παιχνιδιού, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αρχίσει κανείς να μαθαίνει. Βλέπω εδώ στις Βρυξέλλες ε, τόσα πολλά παιδιά που ζουν σε σπίτια που είναι δίγλωσσα. Μέσα στο σπίτι μιλούνται διαφορετικές γλώσσες και τα παιδιά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κάνουν τη διάκριση μεταξύ των γλωσσών που ομιλούνται. Ε, υπάρχει η συμφωνία ε, για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και ξέρουμε ότι το σύστημα εκπαίδευσης, ε, η πολιτική εκπαίδευση είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και πολλά κράτη-μέλη ξέρουμε ότι για την εκμάθηση των γλωσσών πρέπει λίγο να επιταχύνουν την πολιτική τους για να επιτύχουν τους στόχους αυτούς. Και η ερώτησή μου είναι πώς μπορούμε να κάνουμε αυτά τα κράτη-μέλη ε, να τα ενθαρρύνουμε. Δεν μπορούμε να τα υποχρεώσουμε, υποχρεωτικό δεν μπορεί να γίνει, αλλά πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν λίγο τις προσπάθειές τους. και υπάρχουν πολλές ε, μεθοριακές περιοχές. Εγώ είμαι από την περιοχή μεταξύ Ολλανδίας και Γερμανίας και όλοι καταλαβαίνουν και τις δύο γλώσσες. Τουλάχιστον από την πλευρά της Ολλανδίας όλοι ξέρουν γερμανικά. Από την πλευρά της Γερμανίας δεν μαθαίνει κανείς Ολλανδικά. Εδώ χρειάζεται λοιπόν μια δέσμευση. Η δεύτερη γλώσσα θα μπορούσε να είναι η γλώσσα της άμεσα γυτνιάζουσας χώρας. Αυτό διευκολύνει και το να μπορείς να δουλέψεις από την άλλη μεριά των συνόρων. Μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας ίσως είναι λίγο πιο απλό. Μεταξύ Γερμανίας και Ολλανδίας είναι πιο δύσκολο. Μεταξύ Γερμανίας και Τσεχίας ακόμη πιο δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό μοντέλο για να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια πρόοδο. Η γλώσσα είναι πολιτιστική ταυτότητα τη θέλουμε αυτή την πολιτιστική ταυτότητα, θέλουμε και την πολυμορφία και γι' αυτό να προσπαθήσουμε όλα να τα έχουμε διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες για να μπορούμε μέσα σε ένα καθεστώς πολυγλωσσίας να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος από τους δύο θα ήθελε να απαντήσει. Σύντομες απαντήσεις, παρακαλώ. Ο κύριος Στόιτς. Η δεύτερη ξένη γλώσσα σαφώς εξαρτάται από το που ζει ο καθένας και υπάρχουν εξαιρετικά προγράμματα σε διαμεθοριακές περιοχές μεταξύ Γερμανίας, Τσεχίας, παραδείγματο χάρη ή αλλού όλοι θεωρούν σημαντική την εκμάθηση των Αγγλικών και γι' αυτό είναι σημαντικό να προωθούμε την δεύτερη ξένη γλώσσα. Σε, στο τρίγωνο μεταξύ Γερμανίας, Πολωνίας, ε, Τσεχίας ε, είναι διαφορετικές οι γλώσσες από ό,τι μεταξύ Γερμανίας και Ολλανδίας ή μεταξύ Ιταλίας, Γαλλίας, ε, Ελβετίας, παραδείγματος χάρη. Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων έγιναν πολλές εκδηλώσεις σχετικά με το διαμεθοριακό χαρακτήρα της εκμάθησης γλωσσών και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να εξετάσουν τι δυνατότητες υπάρχουν. Υπάρχουν ε, εξαιρετικά προγράμματα για την κατάρτιση των διδασκόντων σε πόλεις όπου ομιλούνται πολλές γλώσσες υπάρχουν πολλές δυνατότητες που προτείνονται και προσπαθούμε να τα υποστηρίζουμε όλα αυτά και μέσω του προγράμματος Εράσμους και θα συνεχίσουμε με εκδηλώσεις όπως αυτές που γνωρίζετε στην Πράγα και αλλού. ένα σύντομο σχόλιο από τη δική μου εμπειρία πριν από 15-20 χρόνια στις εισαγωγικές εξετάσεις αν κάποιο θέλει να, να σπουδάσει κινέζικα ή οποιαδήποτε άλλη ασιατική γλώσσα πρέπει να, γνωρίζει ήδη δύο γλώσσες μία σε υψηλό επίπεδο και μία άλλη που να μπορεί να διαβάζει και να καταλαβαίνει αυτό δεν ισχύει εδώ και πέντε χρόνια όμως αυτή η υποχρέωση διότι η δυνατότητα που έχουν οι φοιτητέ να το κάνουν να, κάνουν απλώ έχει μειωθεί δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Υποτίθεται ότι η κοινωνία μα είναι πιο, όλο και πιο ανοιχτή, οι φοιτητέ έχουν και πιο, όλο και πιο πολλέ δυνατότητε, αλλά μαθαίνουν όλο και λιγότερε γλώσσε. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά σας λέω την εμπειρία μου ως καθηγήτρια πανεπιστημίου στην Πράγα. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην επόμενη συντονίτρια. Παρακαλώ, κυρία που έχετε το λόγο. Merci. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι η ίδια δασκάλα και με ενδιαφέρει το θέμα πολύ. Είμαι καθηγήτρια λοιπόν και είδα αυτό που μας δείξατε, ε, το, τα γραφήματα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί υπάρχουν τόσες μεγάλες διαφορές ε, στις επιδόσεις ε, μεταξύ των χωρών. Δεύτερη ερώτηση. Μήπως, ε, το έλεγε άλλωστε προηγουμένως και η κυρία, ε, ανάμεσα, ε, κάποια σχέση ανάμεσα και στις ελλείψεις των καθηγητών ενδεχομένων που διδάσκουν ξένες γλώσσες. Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε να βρεθεί με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ακριβώς, στη διάρκεια των, της, των σπουδών, ε, να δίνεται η δυνατότητα στους ε, καθηγητές ξένων γλωσσών να πάνε να ζήσουν κάποιο διάστημα στη χώρα της, ε, που μιλιέται η γλώσσα την οποία θα διδάξουν. Πολύ σύντομα. Εγώ έμαθα Κινέζικα στο σχολείο, μια εποχή που δεν μπορούσε κανείς να ταξιδέψει στην Κίνα. Μετά δούλεψα σαν διερμηνέας και Δούλεψα για λίγο και στην Κίνα και τότε με αυτές τις εμπειρίες πραγματικά έμαθα τις γλώσσες, έστω και αν ήμουν πολύ καλή φοιτήτρια εξ αρχής. Νομίζω ότι πραγματικά ε, εάν θέλει κανείς να κατανοεί πραγματικά μια γλώσσα και αν θέλει να κατανοήσει την την πολυπλοκότητα της γλώσσας θα πρέπει οπωσδήποτε να ζήσει σε εκείνη τη χώρα. Αλλά βεβαίως προκύπτει πρόβλημα. Πώς είναι δυνατόν όλο το διδακτικό προσωπικό από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο να έχει την δυνατότητα να ζήσει σε μια άλλη χώρα. Τουλάχιστον για την Τσεχία και τους ε, φοιτητές που σπουδάζουν ε, ξένες γλώσσες, ε, δεν, για να γίνουν καθηγητές ξένων γλωσσών δεν είναι δυνατόν αυτό. Η κυρία Φασόν, παρακαλώ, που είχε ζητήσει το λόγο, αλλά δεν τη βλέπω στην αίθουσα. Δίνω το λόγο, λοιπόν, στην επόμενη ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τις παρουσιάσεις που ήταν και οι δύο πολύ ενδιαφέρουσες. Είμαι σαφώς ε, υπέρ της εκμάθησης ξένων γλωσσών και υπάρχει και ε, χρονικά μια προτίμηση. Όσο νωρίτερα ξεκινήσουν τα παιδιά, τόσο καλύτερα, τόσο πιο εύκολα μαθαίνουν τις ξένες γλώσσες. Η πρώτη γλώσσα είναι τα αγγλικά, ε, η δεύτερη μπορεί να ξεκινήσει ε, και στο σπίτι. Στη Γερμανία από την ε, τρίτη δημοτικού αρχίζει η εκμάθηση των αγγλικών και τη βρίσκω καλή αυτή την προσέγγιση. Τώρα, από την πλευρά της ποιότητας πρέπει να το δούμε σε τι επίπεδο φτάνουν τα παιδιά. θα μπορούσε να βελτιωθεί το επίπεδο, να βελτιωθεί η ποιότητα για να μπορούν πραγματικά να μιλήσουν τα παιδιά που μαθαίνουν τη γλώσσα. Θα πρέπει επίσης να έχουμε και αρκετούς ε, διδάσκοντες, να μην παραμελούμε το διδακτικό προσωπικό. Θα ήθελα να μιλήσω και για το θέμα του ότι η γλώσσα ε, είναι αυτό το οποίο μας φέρνει σε γνωριμία με τον πολιτισμό. Τα συνώνυμα της λέξης πολιτισμού είναι πολλά και ποικίλα. Βλέπω τις εξελίξεις στις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, στα διάφορα πανεπιστήμια με κάποιες δράσεις οι οποίες είναι αντιπαραγωγικές. Και αυτές οι microaggressions που βλέπουμε στα πανεπιστήμια στην Αμερική νομίζω ότι οδηγούν και σε διακριτική μεταχείριση. Δεν βοηθούν την κατανόηση μεταξύ των λαών. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω και προς την κυρία Γεμπού για τις ε, διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Όντως υπάρχουν διαφορές οι οποίες εξηγούνται λόγω των διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων σε κάθε χώρα και λόγω και των ε, μέσων σε άλλες χώρες ξεκινάει πιο γρήγορα η εκμάθηση της ξένης γλώσσας και αυτό είναι ένας παράγον. Υπάρχουν κράτη-μέλη στα οποία υπάρχει ε, μια δεύτερη, αρχίζει να ε, διδάσκεται μια ε, ξένη γλώσσα από την ένατη τάξη και μετά. Η κινητικότητα, το εράσμους που ανέφερε η κυρία Σιόντροβα είναι σημαντικό. Κινητικότητα και των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών μια περίοδος ε, παραμονής στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι πολύ σημαντική. Η καλή παιδαγωγική επίσης. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα για την εκμάθηση των γλωσσών. Δεν είναι εκμάθηση λεξιλογίου ή εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Μπορεί κανείς να μάθει καλύτερα όταν οι παιδαγωγικές μέθοδοι είναι καλύτερες και εξάπτουν το ενδιαφέρον του μαθητού ε, με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών Κινητικότητα λοιπόν, παιδαγωγική. Αυτά είναι παράγοντες που εξηγούν τις διαφορές στην εκμάθηση γλωσσών μεταξύ κρατών μελών και κατάρτιση διδασκόντων. Το αμερικανικό παράδειγμα που αναφέρεται δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να σχολιάσω. Ναι, ακούστε, πιστεύω ότι ο αμερικανικός τρόπος ζωής είναι πολύ διαφορετικός από το δικό μας. Είναι μια διαφορετική κουλτούρα και δίνεται έμφαση ε, στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς είμαστε πιο περίεργοι, έχουμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους άλλους και αυτό δεν είναι κακό. Δίνουμε το λόγο λοιπόν στον επόμενο μιλητή που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δύο λεπτά χρόνου. Ευχαριστώ. Είχε ένα πρόβλημα η συνάδελφος και ανακάστηκε να φύγει. Εξετάσαμε το γράφημα όμως που δείχνει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είναι πολύ πίσω. Η χώρα μου δηλαδή και η χώρα της συναδέλφου. Ε, και αυτό είναι ανησυχητικό γιατί πρόκειται για δύο μεγάλες χώρες πληθυσμιακά. Από την άλλη τα αγγλικά και τα γαλλικά είναι τα πιο οι πιο διαδομένες γλώσσες. Στο γράφημα πάντως φαίνεται ότι πάμε και προς αυτή κατεύθυνση σε σχέση με την περίοδο ε, από το 2003 έως το 2016. Και το όνομα Βασίλειο και η Γαλλία έχουν σημειώσει πρόοδο. Όμως ε, μας είπατε τι γίνεται σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο κάθε χώρας. Τι γίνεται όμως σε επίπεδο περιφερειών. Εγώ ζω στη Βόρεια Αγγλία. Προέρχομαι από το Yorkshire. Και βεβαίω εδώ προφανώ μπαίνει και το θέμα του Brexit. Ε, είναι μοιρασμένη η κατάσταση στην περιοχή μου για το Brexit. Ε, θα ήθελα να ξέρω όμως, ε, ε έχει κάποια σχέση η, το τι έχει ψηφίσει κάποιος ε, με το αν ξέρει γλώσσες, παραδείγματος χάρη. Εγώ πιστεύω ότι ναι αν κάποιο ξέρει, ξέρει μια δεύτερη, μια τρίτη γλώσσα, πιο εύκολα θα ψηφίσει η Remain. Και έρχομαι στο Erasmus Plus τώρα. Εγώ εργάζομαι με νέους ανθρώπους 16-19 ετών και θέλω να τους δώσω τη δυνατότητα να μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη, να ζήσουν μια εμπειρία στην Ευρώπη. Συνήθω τα παιδιά αυτά είναι από την εργατική τάξη. Κοινωνικά είναι χαμηλά. Είναι αυτοί που δεν έχουν τι ευκαιρίε στη ζωή. Θα ήθελα λοιπόν τα ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτέ τι κοινότητε, Διότι αν αυτοί οι νέοι μπορέσουν να ζήσουν μια τέτοια εμπειρία στην Ευρώπη, μπορεί να αλλάξουν και τι νοοτροπίε στη χώρα μα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Ε. Βασίλειο βέβαια. Βλέπουμε μια αύξηση του εθνικισμού και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά ε, τα προγράμματα ε, όπως το Erasmus Plus ε, να φτάσουν σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι και λιγότερο ενταγμένοι στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Έδειξε αυτές τις γραφικές παραστάσεις με τους χάρτες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα σπουδών σε κάθε περιοχή. Δεν έχουμε περισσότερο αναλυτικά στοιχεία για συγκεκριμένες περιφέρειες. Από την αξιολόγηση του Εράσμους ξέρουμε ότι οι συμμετέχοντες έχουν ε, μάθει πάρα πολλά. Έχει βελτιωθεί και, έχουν βελτιωθεί και οι γλωσσικές τους ικανότητες και η κατανόηση της άλλης ε, χώρας. και είναι στο χέρι σας για να προωθήσετε το πρόγραμμα Εράσμου στο μέλλον. Πρόεδρος, ευχαριστώ και δίνουμε τώρα το λόγο στην κυρία Μελμπάντ. θα θέσω το ερώτημά μου στη μητρική μου γλώσσα στα λετωνικά, αφού μιλάμε για πολυγλωσία και γλώσσες. Θέλω να κάνω μια ερώτηση και να μιλήσω από την προοπτική μιας μικρής ε, χώρας με μια μικρή εμβέλειας γλώσσα, γιατί τα λετωνικά σε σχέση με τα γερμανικά, τα αγγλικά ή τα ρωσικά είναι μια μικρή γλώσσα. Η λετονική γλώσσα είναι μια βαλτική γλώσσα. Μια γλώσσα της Βαλτικής, λοιπόν, από την Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια. Και στη χώρα μας διδάσκονται πολλές ξένες γλώσσες στα σχολεία. Πολλές και διαφορετικές, όχι μόνο μία. Μαθαίνουν δύο ή και τρεις. Και ανησυχώ ότι επειδή μαθαίνουν πολλές ξένες γλώσσες, δεν μαθαίνουν σωστά τη λετονική γλώσσα πολλά παιδιά ασχολούνται πάρα πολύ και με τα ψηφιακά μέσα και στον ε, κυβερνοχώρο τα αγγλικά είναι η δεσπόζουσα γλώσσα. Τα παιδιά λοιπόν της Λετωνίας χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους αγγλικά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε τη μητρική μας γλώσσα και να ρωτιέμαι καμιά φορά πόσο καιρό θα μας πάρει μέχρι ότου χαθεί εντελώς η μητρική γλώσσα, γιατί μέσω του ψηφιακού χώρου τα παιδιά μιλούν στην καθημερινότητά τους αγγλικά. Και θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν μελέτες σχετικά με, την, με τον αντίκτυπο που έχει η ψηφιακή εποχή στις μικρές γλώσσες. πιστεύω ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τις μικρές γλώσσες για να διαφυλάξουμε την ε, πολυγλωσία ακόμη και τις πολύ μικρές γλώσσες που μπορεί να μιλούνται από ένα-ενάμιση εκατομμύριο πολίτες. Ευχαριστώ. I to say, and I'm also... Λυπάμαι που λέω, και εγώ μιλάω μια μικρή γλώσσα, ότι οι γλώσσες εξαφανίζονται. Είναι στη φύση της ανθρώπινης ανάπτυξης. Ε, πρέπει να προστατεύσουμε τις γλώσσες μας βέβαια, αλλά μια γλώσσα ζει την φυσική ροή της ζωής της και εξαρτάται από τη χρήση της. Εάν δεν τη χρησιμοποιεί κανείς, αν δεν την καλλιεργεί κανείς, εξαφανίζεται. Και είναι κρίμα. Ε, εμείς ε, διδάσκουμε τηλετονικά στο πανεπιστήμιο, πανεπιστημιακοί ερευνητές ε, προσπαθούν να διαφυλάξουν τις γλώσσες, αλλά οι γλώσσες μπορούν να διαφυλαχθούν μόνο από του ίδιου του ανθρώπου. Εφόσον του ενδιαφέρει πραγματικά η δική τους γλώσσα, την καλλιεργούν και τη χρησιμοποιούν. Έτσι μόνο επιζεί μια γλώσσα. Είναι στο χέρι σας λοιπόν. Έχουμε Άλλο ένα συντονιστή. Έχετε το λόγο, κύριε Κιζιλγιουριακ. Maybe Ίσως είμαι ο μόνος εδώ που δεν μπορεί να μιλήσει τη μητρική του γλώσσα. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω και ούτε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρώπης γιατί είμαι Κύπριος. Θα μιλήσω λοιπόν σε μια άλλη επίσημη γλώσσα της Κύπρου τα ελληνικά. Και θα επανέλθω. Μπορεί να αλλάξω γλώσσα την ώρα που μιλάω. Να μιλήσουμε για ένα κοινό χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν εξασφαλίζουμε ένα κοινό χώρο στην παιδεία και στο πολιτισμό. Και βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς γλώσσες. Όμω εδώ θέλω να προσέχουμε λίγο όταν μιλάμε για πολυγλωσία. Είναι γεγονό ότι κάποιε γλώσσε είναι κυρίαρχε. Και όχι όλε οι γλώσσε έχουν την ίδια αξία και σημασία. Για παράδειγμα, αν κοιτάζουμε στο κόσμο της μετάφρασης, πόσα βιβλία λογοτεχνίας μεταφράζονται από τα μικρά έθνη προς τα αγγλικά, για παράδειγμα, ή στα γαλλικά ή στα γερμανικά, θα δείτε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί ένα κοινό χώρο πολιτισμού στην Ευρώπη δεν γίνεται χωρίς ανταλλαγή μνήμης. Όταν μιλάμε για πολυγλωσία, δεν μιλάμε μόνο για ανάγκη της αγοράς να υπάρχει και ελεύθερη κινητοποίηση των εργαζόμενων για να εργαστούν παντού. Μιλάμε και ουσιαστικά για ένα κοινό πολιτισμικό χώρο. Άρα λοιπόν εδώ επιβάλλεται ανταλλαγή μνήμης, γνωριμία, θα έλεγα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το τι μεταφράζουμε και δεν προσέχουμε πώς μεταφράζουμε. Ακόμα θα έλεγα ότι χρειάζεται και ένα ευρωπαϊκό εκδοτικό οίκο που θα ενισχύσει τις μικρές γλώσσες λογοτεχνία, ποιήση κτλ. για να μεταφραστούν και σε αυτές τις μεγάλες γλώσσες που όλοι μας έχουμε την τάση να, να μάθουμε όπως είναι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά. Ε, επίσης πρέπει να σας πω ότι εμένα στη χώρα μου, στην Κύπρο, and here I want to shift into English to use another language please for translation. Στην Κύπρο υπάρχουν επισήμως δύο γλώσσες και δεν μαθαίνουμε ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Του άλλου. Θα ήταν λοιπόν καλό να υποστηρίζουμε επίσης να μαθαίνει κανείς τη γλώσσα του γείτονά του αυτός που είναι δίπλα μας. Κάτι που δεν το κάνουμε. Δηλαδή μαθαίνουμε μια γλώσσα η οποία ε, μας υπόσχεται πολλά στην αγορά εργασίας. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Ναι, ολοκλήρωσα. Πρόεδρος. Δεν είστε ο μόνος, γιατί και η δική μου μητρική γλώσσα, η γλώσσα των Ρωμά, η ε, Ρωμανέσκη, δεν είναι μία από τις επίσημες γλώσσες, άρα δεν έχω ε, αντίστοιχα διερμηνία. Ε, δεν υπάρχει ε, κάποια απάντηση, οπότε δίνω ένα λεπτό στον κύριο Ρουίς Τεβέσα για την ερώτησή του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. και ευχαριστώ τους ε, εισηγητές που μας μίλησαν για ένα θέμα σήμερα το πρωί πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον. Εγώ προερχόμαι από μια χώρα ε, που δεν έχει μία και μόνη ε, γλώσσα. Ε, και η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας είναι πολύ καλή βέβαια και την υποστηρίζω. Συμβαίνει και στην Ισπανία. Μαθαίνουν ε, βεβαίως ε, Ισπανικά, αλλά ταυτόχρονα μαθαίνουν και μια άλλη γλώσσα, βασκικά, καταλανικά και μετά και τα αγγλικά σαν πρώτη ξένη γλώσσα. Και αυτό πραγματικά αυτό προσθέτει μια, ε, και μια άλλη γλώσσα και συχνά βλέπουμε ότι υπάρχει και άλλη ξένη γλώσσα για ολικά ή γερμανικά. Το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως ακούσαμε, ήδη ε, είναι υπερφορτωμένο με την εκμάθηση γλωσσών. Υπάρχουν τέρασμος πλάσα, αλλά υπάρχουν και άλλα. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που αποτελεί ευκαιρία ε, για τους νέους να μάθουν και μία άλλη ε, ξένη γλώσσα και μάλιστα κάποια που ενδεχομένως δεν έχουν καταφέρει να σπουδάσουν ε, στο εκπαιδευτικό σύστημα μπορούν επομένως στα πλαίσια του σώματος αυτού να μετακινηθούν, να ζήσουν σε μια άλλη χώρα και να μάθουν από το μηδέν μια ξένη γλώσσα. Ich würde gern die Fragen alle zusammenfassen, damit wir δεν έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να συνεχίσουμε και γι' αυτό θα πρέπει να πάρουμε όλες τις ερωτήσεις μαζί και να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κυρία Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στον εκπρόσωπο της Επιτροπής ήθελα να ε, κάνω μια ερώτηση και στη συνέχεια των όσων ε, είπε προηγουμένως ο Ισπανός συνάδελφος. Έχουμε στην Ισπανία μεγάλη παράδοση γλωσσών. Όμως ε, θέλω να καταγγείλω ότι ε, σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας δεν δίνεται η δυνατότητα να μάθουν τη γλώσσα της χώρας, τα ισπανικά, δηλαδή στις Βαλερίδες νήσους, καθώς επίσης και στην Καταλωνία υπάρχουν περιοχές όπου τα παιδιά δεν έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν στην μητρική τους γλώσσα. Και από τη στιγμή που μιλάμε για την Ευρώπη, για το πολιτιστικό της αγαθό, για την πολιτιστική της περιουσία, ε, ε, ε, θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν την δυνατότητα να διδαχθούν στη γλώσσα των γονιών τους, στη μητρική τους γλώσσα. Θα πρέπει στην Ισπανία λοιπόν τα παιδιά να έχουν την δυνατότητα να μάθουν τα Ισπανικά. Μετά να τους δίνεται βεβαίως η δυνατότητα, η εξαιρετική δυνατότητα να μαθαίνουν μαθαίνουν και άλλες γλώσσες. Αλλά τονίζω και καταγγέλω ότι υπάρχουν ε, παιδιά τα οποία δεν έχουν αυτή τη στιγμή στην Ισπανία το δικαίωμα να εκπαιδευτούν, να διδαχτούν την μητρική τους γλώσσα. Κύριε Μπόσκο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω μετά από αυτό που προηγούμενος ομιλητής ότι δεν, και να πω ότι δεν είναι μόνο σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε ε, ε, να μαθαίνουμε, να εκπαιδευόμαστε στη δική μας γλώσσα και στη γλώσσα τη μητρική ανθρώπων που προέρχονται από μειονότητες πρέπει και άνθρωποι που ζουν στη χώρα να μάθουν τη γλώσσα της μειονότητας διότι ε, αυτό θα διευκολύνει και την συμβίωση Τα προγράμματα Εράσμους βοηθούν τους φοιτητές να βελτιώσουν τις γλώσσες τους και την προφορά τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να προσελκύσουμε ε, βεβαίως και ομιλητές ε, που μιλούν τη μητρική τους γλώσσα ε, για να μπορούν οι φοιτητές να μαθαίνουν ε, να μαθαίνουν σωστά τη γλώσσα. Ορισμένε φορέ δηλαδή πρέπει να μετακινείται ο καθηγητή, όχι απαραίτητα οι φοιτητέ μόνο. Ο κύριος Σέρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Από τη Σλοβενία έρχομαι και τα σλοβενικά τα μιλούν περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Είναι θαύμα το ότι η γλώσσα μας έχει επιβιώσει. Η χώρα μας είναι μεταξύ της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Γερμανίας, άλλων σλαβικών χωρών πολλές, πολλές μεγάλες δηλαδή ε, γλωσσικές ε, ενότητες μας ε, περιτριγυρίζουν, αλλά διαφυλάξαμε τη, χώρα, τη γλώσσα μας γιατί διαφυλάξαμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα για αιώνες. Ε, γι' αυτό παρέμεινε η γλώσσα μας τόσο ισχυρή. Τώρα, είναι πολύ ενδιαφέρον το γράφημα που μας παρουσιάσατε για τις δεξιότητες, τις γλωσσικές, για την πρώτη ξένη γλώσσα. Είναι αλήθεια ότι οι μικρές χώρες είναι οι πιο επιτυχείς, διότι είναι υποχρεωμένοι να μάθουν τις γλώσσες των μεγάλων χωρών. Αυτή είναι η απάντηση. Παρακαλώ, επόμενος ομιλητής. Η κυρία Γκριζέ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην πολυγλωσσία ε, από ένα πιο πολιτικό πρίσμα και να θέσω ένα ερώτημα στην Κομισιόν. Σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Μέρα των Γλωσσών δεν υπάρχει κάτι το παράδοξο όταν εδώ ηγεμονεύουν τα αγγλικά. Ο κάθε βουλευτή θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα κοινοβουλευτικά έγγραφα στην επίσημη γλώσσα που προτιμά. Και αυτό ε, δεν μπορεί να το έχει ε, και είναι κάτι που παραβιάζει τα δικαιώματά του να το λέει, ε, το λέει η νομολογία. μιλάμε το το 158 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Μιλάμε για το καθεστώ των Ευρωπαίων, των, των Ευρωβουλευτών, που λέει ότι όλα τα έγγραφα του Κοινοβουλίου πρέπει να ε, συγγράφονται ε, σε όλες τις γλώσσες. Η, η διαμεσολαβήτρια είπε ότι πρέπει να έχει κάνει πρόσβαση σε, έγγραφα, ε, ο πολίτης να έχει πρόσβαση σε έγγραφα στη γλώσσα που να γνωρίζει. Διότι αυτό, αυτό δημιουργεί μεγάλη επιφυλακτικότητα. Πρέπει οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να ασκήσουν το, το δημοκρατικό του δικαίωμα του ελέγχου. Πώ θα διασφαλίσουμε σε όλου του βουλευτέ ότι θα σεβαστούν τα εκπροσωπικά του δικαιώματα και να υποχρεώσουμε θεσμικά όργανα ε, να σεβαστούν τι υποχρεώσει που έχουν αναλάβει. Ευχαριστώ. Κύριε Τόιτς, νομίζω θα θέλετε να απαντήσετε. Όταν μιλάμε για την γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη, μιλάμε για όλες τις ε, γλώσσες, και τις εθνικές αλλά και τις περιφερειακές γλώσσες. Και υπάρχουν πολλά προγράμματα στο πλαίσιο του Εράσμους ε, που προωθούν και τις ε, μικρές γλώσσες. Στο Ευρωπαϊκό Έτος ε, Γλωσσών είχαμε πολύ καλά προγράμματα για την εκμάθηση πολλών γλωσσών συμπεριλαμβανομένων και των περιφερειακών γλωσσών και στη Βαλένσια και ε, στην Καταλονία είχαμε ένα πολύ καλό έργο και στη χώρα των Βάσκων. Προωθούμε δηλαδή όλες τις γλώσσες, προωθούμε και τις μικρές γλώσσες. και είναι σημαντικό και για τους διδάσκοντες, όπως ε, είπε μια ομιλήτρια. Ε, στο πλαίσιο του Εράσμους προωθούμε και την ε, κατάρτιση των διδασκόντων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Λόμοβα και κύριε Τόιτς για τις παρουσιάσεις σας. Ευχαριστώ και τους συντονιστές. Σας αποχαιρετίζουμε λοιπόν. Σας αποχαιρετούμε τους προσκεκλημένους μας και συνεχίζουμε σε μια συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης. Έχουμε μια συζήτηση στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης, για την οποία καλωσορίζω το Διευθυντή του Κέντρου Μετάφρασης, τον κύριο Μπενουά Βιτάλ. Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι αξιότιμοι βουλευτές, σε αυτήν τη βδομάδα ε, όπου υπάρχει η μέρα των Ευρωπαϊκών Γλωσσών μετά από μια γενική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετάφρασης, του Κέντρου Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Γλωσσών, εν πάση περιπτώσει, Παρακαλώ, διακόπτει ο πρόεδρο. Ε, ήσυχα όσοι αποχωρούν από την αίθουσα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Έλεγα λοιπόν ότι μετά από μια γενική παρουσίαση του Κέντρου Μετάφραση των Οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα ε, για την περίοδο 2018 θα σα ε, μιλήσω για τα, ε, τις, τα θετικά στοιχεία, τα αρνητικά, τι δυνατότητε που υπάρχουν. Πριν από 25 χρόνια δημιουργήθηκε αυτό το κέντρο ε, η βάση του είναι στο Λουξεμβούργο έχει τις δικές του, του οικονομικούς πόρους που προέρχονται αποκλειστικά από την πληρωμή των υπηρεσιών προς τους πελάτες του. Δηλαδή δεν έχει οποιαδήποτε άλλη επιδότηση. Το 2018 το κέντρο βασιζόταν σε 183 υπαλλήλους και 23 προσωρινούς υπαλλήλους. Υπάρχει ένας γενικός διευθυντής και, και ένα διοικητικό συμβούλιο. Εδώ βλέπετε το οργανόγραμμα. Ε, το οποίο βασίζεται σε τέσσερις ε, ε διευθύνσεις με 100 περίπου μεταφραστές που μεταφράζουν στις 24 γλώσσες. Γιατί το κέντρο μεταφράσεων δημιουργήθηκε από την Ευρωπαίο νομοθέτη. Λέει ο κανονισμός, λέει ο κανονισμός ότι το κέντρο θα εξασφαλίσει τις υπηρεσίες μετάφρασης που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των οργανισμών και είναι το μοναδικό εξειδικευμένο κέντρο που καλύπτει τις ανάγκες μετάφρασης σημαντικού αριθμού θεσμικών οργάνων που είναι διασκορπισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα έχοντας κατά, μέτω, κατά ε, νου το, την ορθολογική διαχείριση. Θέλουμε να κάνουμε προφανώς ε, οικονομίες κλίμακας, μιας και είναι πολλές, ε, πολλοί συνδυασμοί γλωσσών, ε, να μην δημιουργηθούν μήνυ υπηρεσίες μετάφρασης, ε, ε, να μην ξεκινήσουν πολλαπλοί διαγωνισμοί. Ποιος, ποια είναι η αποστολή του κέντρου μετάφρασης. Είναι πολλαπλή. Αφενός θέλουμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επικοινωνήσουν στη γλώσσα όλων των πολιτών και να μεταφράσουμε βεβαίως και να δώσουμε άλλες υπηρεσίες, να παράσχουμε άλλες υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφραστικές που χρειάζονται ε, οι ε, πελάτες μας, χρησιμοποιώντας βεβαίως τις, και τις νέες τεχνολογίες, ε, δημιουργώντας ε, τις, την κατάλληλη προσφορά υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 67 πελάτες για μας, όργανα ε, και ε, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως έχουμε και νέες όπως το Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Κάποια αριθμητικά στοιχεία τώρα σημαντικά. Το κέντρο έχει ένα προπολογισμό περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ. Το 2018 ήταν 41,2 εκατομμύρια ε, τα έσοδα, 44 ε, εκατομμύρια τα έξοδα, 3 εκατομμύρια έλλειμμα δηλαδή, που καλύφθηκε από ένα απόθεμα που υπάρχει, απόθεμα για την σταθερότητα των τιμών, έτσι λέγεται. 369.000 σελίδες μεταφράσεων, 412.000 ε, ευρωπαϊκών σημάτων, 672 ε, ημέρες ε, εργασίας. Βασιζόμαστε στην εξωτερική μετάφραση και βεβαίως υπήρξαν σημαντικές διορθώσεις γλωσσικές αυτές τις εξωτερικές μεταφράσεις. Η μέση τιμή ανασελίδα για τους πελάτες μας είναι 68 ευρώ 16% δηλαδή από το στάνταρ τιμές διότι η πολιτική μας λαμβάνει υπόψη της τη χρήση ε, των, της μνήμης μετάφρασης που υπάρχει για να μειώσει το κόστος. Βλέπετε εδώ τον αριθμό των σελίδων που ε, μεταφράστηκαν με τον καιρό. Αυτό έχει να κάνει και με τη διεύρυνση, μεγάλη αύξηση. Προσαρμόσαμε προφανώς και εμείς το προσωπικό μας ε, με βάση τις ανάγκες από το 2010 το προσωπικό βεβαίως έχει αρχίσει να μειώνεται από 2015 είμαστε 183 πλέον μόνιμοι υπάλληλοι ή προσωρινοί υπάλληλοι 193 ε, προβλέπονται για το 2018 υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία όπως βλέπετε σε ό,τι αφορά τους πελάτες μας και υπάρχει και μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά τον όγκο εργασίας είναι πολύ μικροί πελάτες που χρειάζονται τις υπηρεσίες μας και που δύσκολα θα μπορούσαν να απευθυνθούν στην ιδιωτική αγορά ε, για να βρουν τις υπηρεσίες που τους προσφέρουμε εμείς. Εδώ τώρα νομίζω ότι θα προσφέρει ενδιαφέρον αυτό το, αυτή η διαφάνεια για την Αντιπρόεδρο. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι τα αγγλικά ως γλώσσα πηγής εκπροσωπεί 90% αποτελεί 90% των κειμένων που μεταφράζονται. Έτσι. Ε, δυστυχώς δεν φαίνεται εδώ καν τα λετωνικά είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Πολύ κάτω από το 1%. Επίσης μεταφράζουμε και προς κάποιες μη ευρωπαϊκές γλώσσες 3% περίπου 11.769.000 σελίδες. Κάποια, σελίδες, κάποια λόγια τώρα για, την, για το οικονομικό μοντέλο. Είπαμε ότι τα έσοδά μας προέρχονται αποκλειστικά από τα, τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και τις σχετικά τιμολόγια υπάρχει ανάθεση 86% της παραγωγής μας προς εξειδικευμένους μεταφραστές, περίπου ένα τέταρτο προπολογισμού μας, 11 εκατομμύρια του χρόνου περίπου. Αυτές οι μεταφράσεις βεβαίως στη συνέχεια 100% ελέγχονται σε ιστορικό επίπεδο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε 24 γλωσσικές ομάδες. Έχουμε μικρές ομάδες μετάφρασης, που εξασφαλίζει τις επίγουσες ή τις ε, εμπιστευτικές μεταφράσεις και όπως σας είπα ε, προφανώς επαληθεύουμε την ορθότητα των μεταφράσεων που έχουν ανατεθεί εκτός ε, της υπηρεσία μας. Βασιζόμαστε πλέον και στην αυτόματη μετάφραση και στις ε, βάσεις δεδομένων, δηλαδή ε, λιμάτων. Αυτά χρησιμοποιούνται πλέον συστηματικά εργαζόμαστε σε πολλού και διάφορου τομεί, διότι οι υπηρεσίε μα είναι ευρωπαϊκέ ε, υπηρεσίε. Οι πελάτε μα είναι ευρωπαϊκέ υπηρεσίε. Μπορεί να είναι ο οργανισμό φαρμάκου, διατροφική ασφάλεια, σιδηρόδρομοι, αερομεταφορέ ε, και βεβαίω υπάρχει πλέον και οι ε, η τραπεζικοί οργανισμοί. Η βασική υπηρεσία μα είναι η μετάφραση, η δουλειά που γίνεται σε παιδορολογία. Προσπαθούμε η μετάφραση να είναι όσο γίνεται πιο εύκολη ε, και για τις ιστοσελίδες, ε, διότι είναι ο τομέας όπου χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Ε, υπάρχει μια διαδικασία εξασφάλισης της ποιότητας, αυτή είναι η προσθέμενη αξία μας. Αυτό έχει να κάνει και σε ό,τι αφορά τα κριτήρια πρόσληψης και σε ό,τι αφορά την διαβίου μάθηση και βεβαίως όταν εξωτερικοί συνεργάτες ε, δεν είναι ποιοτικοί αποκλείονται ε, υπάρχει μια σημαντική προπαρασκευή και μια παρακολούθηση ε, προσπαθούμε να μετρήσουμε και το επίπεδο ικανοποίηση των πελατών μας το κέντρο εξασφαλίζει την διαχείριση της μεγαλύτερης βάσης δεδομένων παγκοσμίω σε, πεδρολογία. Τώρα, ποια είναι ε, τα θετικά και τα αρνητικά σημεία, οι δυνάμεις και τα δυνατά σημεία και αυτές αδυναμίες. Ε, το κέντρο διευκολύνει την πολιτική της πολυγλωσσίας. Ε, έχει δημιουργήσει μια οργάνωση και εργασίες και εργαλεία αποδοτικά διαχείρισης της δραστηριότητα. Έχουν ελεγχθεί αρχές 2019 από τις υπηρεσίες ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έφτασε στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία και τα εργαλεία είναι κατάλληλα, είναι αποτελεσματικά και λειτουργούν. Αυτό περιμέναμε και εμείς. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της οργάνωσης είναι ε, μια έντονη αυτοματοποίηση των καθηκόντων που βασίζεται σε αλγόριθμους εστιασμένους και συστηματική χρήση μνήμης μετάφρασης. Ε, η αυτόματη μετάφραση χρησιμοποιείται, όπως είπα, ε, όλο και περισσότερο. Λοιπόν, τώρα, ποιες είναι οι αδυναμίες μας. οι πελάτες έχουν την εντύπωση ότι πληρώνουν ακριβά για μια υπηρεσία μετάφρασης ε, για την οποία έχουν την εντύπωση ότι θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση δωρεάν μέσω Google, Deeple ή Translation κτλ. Ε, έχει σημαντικά διαστρωτικά, διαστρωτικό κόστος, βρίσκεται στο Λουξεμβούργο το κέντρο αυτό, ε, πρέπει να σεβαστούμε το καθεστώς των υπαλλήλων και το, υπάρχει και οικονομικός κανονισμός, υπάρχει υποχρέωση ισότιμης ε, μεταχείρισης όλων των γλωσσών, ε, κάτι που δεν συμβαίνει εκτός ε, στην, στην ιδιωτική αγορά, ο κίνδυνος είναι ότι οι πελάτες μπορεί να θελήσουν να απευθυνθούν αλλού για αυτές τις γλωσσικές υπηρεσίες, ε, ερμηνεύοντας τον υπάρχοντα κανονισμό που λέει ότι οι υπηρεσίες μετάφρασης είναι, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία. Οι υπηρεσίες μετάφρασης λέμε έτσι, εάν το ερμηνεύσουμε αυτό ευρέως ε, θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε θα μπορούσε να οδηγήσει ότι ε, με την άφηξη της τεχνητής νοημοσύνης ε, και θεωρήσουμε ότι η κλασική διαδικασία προετοιμασία, αυτόματη μετάφραση και επανεξέταση φεύγει η λέξη μετάφραση. Ε, δηλαδή θα μπορείς ο πελάτης να ερμηνεύσει τον κανονισμό και να πει ακούστε υπάρχουν μηχανήματα που μεταφράζουν ε, δεν είναι μετάφραση αυτό χρησιμοποιώ αυτά τα μηχανήματα και απευθύνω εξωτερικό συνεργάτη και για την επαλήθευση στη συνέχεια χωρίς να περνάω από το κέντρο τι γίνεται στην περίπτωση αυτή ε, δώστε μου ένα λεπτό ακόμα πρόεδρε πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Υπάρχει και ένα σχέδιο ε, κάποιων μετατροπών. Θέλουμε να τα πάμε πιο κοντά στους πελάτες μας με τις υπηρεσίες μας. Πρέπει να πάμε όμως ακόμα παραπέρα. Και εδώ έχουμε δύο εναλλακτικέ αυτή τη στιγμή που προετοιμάζουμε. Να καθορίσουμε σαφέστερα την υπηρεσία μετάφρασης, είναι γλωσσική υπηρεσία ε, γραπτή και θέλουμε να αντικαταστήσουμε το κείμενο υπηρεσίες μετάφρασης από τον όρο γλωσσικές υπηρεσίες στο γραπτό τομέα, γραπτός. Τα κλασικά κείμενα που παρουσιάζονται, που αναφέρονται στους κανονισμούς των νέων υπηρεσιών και ε, στους ε, υπάρχοντες κανονισμούς που δημιουργούν διάφορους ε, ε, δημιουργίες των διαφορών ε, υπηρεσιών, όλα αυτά να αναφέρουν αυτή τη διατύπωση. είπαμε ότι είναι πάρα πολλοί γλωσσικοί συνδυασμοί. είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να δίνουμε στην, στο, κέντρο αυτό τα μέσα που χρειάζεται για να συνεχίσει να διευκολύνει τους πελάτες να μπορούν οι, πελά, οι αυτοί να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική πολυγλωσσίας όπως είπατε και εσείς Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια επιστολή που στείλατε στον πρόεδρο του κέντρου το 2018. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βιτάλ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε καθόλου χρόνο όπως βλέπετε. Δεν θα έχουμε διερμηνήσει μετά από λίγο. Έχουμε πολύ σύντομο χρόνο για πιθανές ερωτήσεις. Αλλά να είστε πολύ σύντομοι στις ερωτήσεις σας. Μπορώ να κρατήσω ένα κατάλογο μιλητών. Ποιο θα ήθελε το λόγο. Δεν βλέπω να θέλει κανείς το λόγο. Α, παρακαλώ. Ο κύριο Λάμποκοφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Βιτάλε, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή Λέτε ότι η αποστολή σας είναι να βοηθήσετε τις, ε, ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσον αφορά τα θέματα μετάφρασης και από ό,τι καταλαβαίνω δουλεύετε πολύ, συνεργάζεστε με πολλές ε, υπηρεσίες, οργανισμούς ευρωπαϊκούς και υπογραμμίζετε το θέμα της ποιότητας. και ότι εντάσσεστε κατά αυτή την έννοια στην προσπάθεια πολυγλωσσίας και πρόθεσης της πολυγλωσίας στην Ευρώπη. Ε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προτείνετε και ε, ε, μεταφράσει σε άλλες γλώσσες. Η ερώτηση μου είναι ποιες είναι οι άλλες γλώσσες, ποιες είναι αυτές οι άλλες γλώσσες, ποιο είναι το ποσοστό των μεταφράσεων σε αυτές τις, προς αυτές τις γλώσσες. Ε, η πολιτική μου ομάδα μου έχει αναθέσει να μελετήσω ε, το θέμα αυτό ε, και στα πλαίσια της, του ελέγχου του προϋπολογισμού. Γι' αυτό θα ήθελα αυτές τις, τα στοιχεία από σας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη εμιλήτρια, ένα σχόλιο και μια ερώτηση. Όταν μεταφράζεται για το Κοινοβούλιο, καλό θα ήταν να χρησιμοποιείτε πάντα τις ε, ίδιες ε, ε, συντομεύσεις για τις πολιτικές ομάδες. Είμαστε 600 νέοι βουλευτές. Όταν ας πούμε γράφετε PPE να ξέρουμε ότι παντού θα είναι το ίδιο. Επίσης, ε, είσαστε προετοιμασμένοι ή έχετε πρόθεση να χρησιμοποιήσετε, να κάνετε μεταφράσεις ας πούμε προς την νοηματική. Δηλαδή, εάν ε, εάν υπάρχει κάποιος ε, κοφός ο οποίος προέρχεται από οποιαδήποτε χώρα. Ο κύριος Βιτάλη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο ρόλος ε, του κέντρου είναι να μεταφράζει, μετάφραση των κειμένων λοιπόν. Ε, επομένως δεν μπορεί δυστυχώς να ασχοληθεί με την νοηματική, τουλάχιστον όχι σήμερα. Δεν ξέρω αν αργότερα θα έχει την δυνατότητα αυτή, αν θα ασχοληθεί με αυτό. Πάντως προς ώρας ε, δεν αποτελεί αρμοδιότητά του. Ε, αναφέρεστε φαντάζομαι στην διερμηνία στην νοηματική γλώσσα. Ε, ε, όχι, δεν υπάρχει μετάφραση, πρέπει να μιλήσουμε για διερμηνία. weiteren Fragen. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη ερώτηση. Οπότε κλείνουμε τη συνεδρίαση, αγαπητοί συνάδελφοι, και θα τα ξαναπούμε στις 3 για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Καλό σας μεσημέρι.